ποίησης. Τον λόγο έχει ο εισηγητής μας για τέσσερα λεπτά. Πάνε Πρεσεράιτσι, Βάζενα Κομίσε, Βάζενα... Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Αγαπητοί συνάδελφοι, η έκθεση που θα συζητήσουμε σήμερα έχει υποβληθεί σαν προπομπός του πακέτου τυποποίησης της Κομισιόν. Αυτό το πακέτο θα αναθεωρήσει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο της τυποποίησης, θα την προωθήσει δε μελλοντικά. Γι' αυτό θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα προς την Κομισιόν και προς το κοινό ευρύτερα όσον αφορά την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής τυποποίησης. Ένα αποτελεσματικό σύστημα είναι κλειδί στο επίκεντρο των εξελίξεων για την εσωτερική αγορά και για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας. Γι' αυτό έχουμε αποδώσει ιδιαίτερα προσοχή, ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το θέμα. Είχαμε έντονες συζητήσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους στο πανευρωπαϊκό επίπεδο και με τα κράτη-μέλη. Αναζητούμε λοιπόν ένα μέγιστο σύστημα τυποποίησης. Δεν έχουμε ξεχάσει και τους εκπροσώπους των μικρομεσαίων καθώς και τους καταναλωτές και τα άτομα με ειδικέ ανάγκες και τους περιβαλλοντολόγους. Κανένα δεν έχουμε αφησίαξει. Λοιπόν, συζητώντας αυτό το σύστημα καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η αναθεώρηση δεν πρέπει να οδηγήσει σε ριζικές αλλαγές που θα υπονομεύσουν τον πυρήνα του υφιστάμενου ε, συστήματος. Για να είναι αποτελεσματικό το σύστημα πρέπει οι εθνικοί φορείς που μέχρι σήμερα δεν ήταν ιδιαίτερα ε, ενεργοί να δραστηριοποιηθούν περισσότερο. Οι φορείς τυποποίησης, οι εθνικοί φορείς τυποποίησης ε, είναι η βάση αν θέλετε, τα θεμέλια της ευρωπαϊκής τυποποίησης. Μελλοντικά λοιπόν ακόμη θα πρέπει να καλούμε τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν περισσότερο στη διαδικασία τυποποίησης. Θέλουμε να είναι πιο αντιπροσωπευ... αντιπροσωπευτικός ο μηχανισμός. Προσβασιμότητα τώρα στα πρότυπα αυτά. Τα πρότυπα πάντα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των χρηστών. Πρέπει να είναι φιλικά προς τον χρήστη. Με την απελευθέρωση των υπηρεσιών πρέπει να σκεφτούμε και την τυποποίηση των υπηρεσιών. Είναι κλειδί οι υπηρεσίες για τον διασυνοριακό ανταγωνισμό. Με τον τρόπο αυτό θα καταργήσουμε φραγμούς στην εσωτερική αγορά. Καταργώντας τα εμπόδια και τους φραγμούς θα προχωρήσουμε. Ακόμη θα εξασφαλίσουμε καλύτερο ανταγωνισμό και έτσι διαφάνεια και καλύτερη ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Καινοτομία τώρα και νέες τεχνολογίες. Προωθητικός παράγων αυτός. Άρα χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών ερευνητών και καινοτόμων. Χωρίς αυτή τη συνεργασία η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να τυποποιήσει τις γνώσεις της παραδείγματος χάρη στην ανοτεχνολογία, στην τεχνολογία της πληροφορίας κτλ. Δεν μπορούμε πάντα να μεταφράζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας στην πρακτική. Αν τα καταφέρουμε καλύτερα θα παίξουμε ρόλο κλειδί ευρύτερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους από την Επιτροπή μου και την Επιτροπή Έτρα που με βοήθησαν να συντάξω αυτή την έκθεση. Χαίρομαι που καταλήξαμε σε συμφωνία μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων. Ε, η κυρία Κόμη λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την εργασία και συνεργασία με τον εισηγητή και με τους άλλους σκιώδεις για να βρούμε, να φτάσουμε σε μια σωστή εξισορρόπηση μεταξύ των διαφόρων πολιτικών θέσεων. Έτσι, αποστέλουμε ένα ουσιώδες μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μελλοντική αναθεώρηση. Το παρόν σύστημα λειτουργεί καλά και δεν χρειάζεται ριζοσπαστικές αλλαγές. Οι αλλαγές που προτείνουμε δεν ε, προδικάζουν, μάλλον δεν αλλάζουν την ουσία του υπάρχοντος συστήματος. Γι' αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα, μια νέα τυποποίηση λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα της ΜΜΕ μέσα στα πλαίσια της τυποποίησης. Αυτή δεν είναι παρά η απαρχή και τους επόμενους μήνες θα εργαστούμε στεναρά έτσι ώστε να επιβάλλουμε μια νέα τυποποίηση πανευρωπαϊκά. Ε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ το συνάδελφο που ε, προετοίμασε αυτή την ε, σημαντική έκθεση η τυποποίηση είναι ύψης της σημασίας για την προώθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την άρση των εμποδίων προς το εμπόριο. Ελπίζω να είναι αρκετά εκτενές το πλαίσιο για να καλύψει τις ελλείψεις ως προς την προστασία των προϊόντων. Τα ενιαία πρότυπα διακοινωτικά είναι ύψης της σημασίας για την τεχνολογία και την καινοτομία, για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την υγεία των πολιτών μας, θέτοντας ασφαλή προϊόντα στην αγορά. Ο κύριος Πάσκα, για ένα λεπτό. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης είναι τμήμα του Διεθνού Συστήματος Τυποποίησης. Εδώ ορίζονται οι διεθνείς προδιαγραφές. Η κοινωνία μας μεταβάλλεται ταχύτατα καθώς και ο τρόπος ε, διαβίωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα και να προσαρμοστούν ανάλογα η τυποποίηση. Θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτη και πιο ανοιχτή. Εάν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να είναι πετυχημένη, θέλουμε να έχουμε μια οικονομία η οποία λειτουργεί καλά. Άρα χρειαζόμαστε νέους κανόνες, μια καινούρια τυποποίηση, ούτως ώστε να μπορούν τα νέα προϊόντα να φτάνουν στην αγορά έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου ή να ανανεωθούν οι μηχανισμοί της ευρωπαϊκής τυποποίησης και να αναθεωρηθούν. Μέχρι στιγμής βασίζονται σε εθνικές παραδόσεις. Δεν έχουν εξυγχρονιστεί και θα πρέπει να εξυγχρονιστούν και να προστευθούν. Eh, Κύριε Πρόεδρε, εμείς ως εκπρόσωποι της ε, ΙΟΠΙΚ ε, χαρακτηριζόμαστε πολύ συχνά ως ευρωσκεπτικιστές. Είμαστε πράγματι ευρωσκεπτικιστές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε να υποστηρίξουμε τη συνεργασία μεταξύ των χωρών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε κατά της βασικής αρχής να γίνουμε οι Ηνωμένε Πολιτείε της Ευρώπης. Ωστόσο το ζήτημα της τυποποίησης ε, θέλουμε να το στηρίξουμε. Όλοι μας επικρίνουν και μας λένε ότι παλεύουμε εναντίον των πάντων. Δεν είναι αλήθεια. Εμεί θέλουμε να προωθηθεί αυτό το θέμα. Στηρίζουμε το θέμα της τυποποίηση και θέλουμε πραγματικά να σας παρακαλέσουμε να δώσετε, να παράσετε και τη δική σας υποστήριξη και να υπερψηφίσετε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω δύο ακόμα μιλητές. Πρώτα η κυρία Μπασέσκου για ένα λεπτό. Η προώθηση του ευρωπαϊκού πλαισίου τυποποίησης μπορεί να βοηθήσει την θέση των ΜΜΕ τα ΜΜΕ χρειάζονται αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης έτσι ώστε να μην υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία καθώς και ένα απλό σύστημα χρηματοδότησης. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης θα πρέπει να προωθήσει την καινοτομία και να αποτελέσει κοινή βάση για την περαιτέρω τυποποίηση. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να ισχύει η αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Γι' αυτό το, Think Small First θα πρέπει να ισχύει και για τις ΜΜΕ. Επίσης θα πρέπει να πω ότι στη Ρουμανία πρόσφατα προβλέπονται μέτρα για την εφαρμογή της νομοθεσίας ΕΕ μέσα στα πλαίσια μια κοινή βάση ε, τυποποίησης. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση αποστέλει ένα άλλο μήνυμα στην Επιτροπή για να συνεχίσει με την εναρμόνιση των προδιαγραφών και προτύπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να υπερασπιστούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι των, των προϊόντων χαμηλής ποιότητας που προέρχονται από την Ασία. Θα σας... Ήθελα να σας ευχαριστήσω διότι υποστήριξα την τροποποίησή μου για να υπάρχουν ασφαλή υποδήματα για τα παιδιά. Δυστυχώς πολλά παιδιά έχουν μεγάλα προβλήματα στα πόδια εξαιτίας των κινέζικων υποδημάτων που κυκλοφορούν. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν ασφαλή προϊόντα και αυτό αφορά και τα υποδήματα αλλά και τα παιχνίδια. Ελπίζω η Επιτροπή να ανταποκριθεί σε αυτή την ε, πρόκληση γιατί Δυστυχώς το λόμπι της Γαλλίας και της Γερμανίας προβάλλουν ε, μία συστηματική θέση έτσι ώστε να μην έχουμε μία ενιαία φωνή. Ε, Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Είναι μία πολύ καλή αρχή για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης και τη στιγμή που μιλάμε για τις πιο ευπαθείς ομάδες, τους καταναλωτές, τους οικολόγους, όλοι αυτοί οι φορείς θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στην τυποποίηση. Δεν θα πρέπει να είναι μόνο το γήπεδο παιχνιδιού των μεγάλων επιχειρήσεων, της big business. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την σωστή εκπροσώπηση όλων των ομάδων συμφερόντων. Όλοι θα πρέπει να εισακουστούν. Επίσης, αυτές οι ομάδες συμφερόντων θα πρέπει να ενισχυθούν. Νομίζω ότι μπορούμε να ενισχύσουμε τον ρόλο τους ε, εάν έχουν δικαίωμα ψήφου στις τεχνικές επιτροπές. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε και μία δεύτερη γραμμή παραγωγής και ελπίζω αυτό να το... Καληνύχτα σας. Ευχαριστώ πολύ όλους που χρησιμοποίησαν ελληνικά και, και με κάνουν να μην αισθάνομαι τόσο μόνος στην, στη βραδινή βάρδια του, της Ολομέλειας. Ε, και αυτό αφορά και την τελευταία ομιλήτρια για την ημέρα, την ε, κυρία Δαμανάκη, εξ ονόματος της Επιτροπής. like to Θα ήθελα να συγχαρώ τον ε, εισηγητή για την ε, περιεκτική του έκθεση η οποία χαίρει της γενικής αποδοχής. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου που έμειναν εδώ μέχρι αργά για να βοηθήσουν τον πρόεδρο στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του και να προβάλλουν κάποιε πολύ επικοδομητικέ και χρήσιμε ιδέε στη συζήτηση. Αυτή η έκθεση είναι μια σημαντική συνεισφορά στη συζήτηση που άρχισε πριν από μερικά χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μα ευστά την προσοχή όσον αφορά το μέλλον του συστήματο τυποποίηση στην Ευρώπη, ένα κεντρικό στοιχείο στην εφαρμογή τη εσωτερική αγορά, στην αύξηση τη ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και ένα σημαντικό εργαλείο για τη διευκόλυνση των καινοτομιών. Ε, στην επικείμενη συζήτηση η ευρωπαϊκή τυποποίηση θα πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες ενεργειακές, ε, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις, όπως ήδη αναφέρεται. Υπάρχει μεγάλη, υπάρχουν νέες αναδυόμενες οικονομικές ε, δυνάμεις, διαχείριση του άνθρακα, κλιματικές προκλήσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όλα αυτά είναι διάφοροι παράγοντες που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε παρόλο που παρόλο και αν τα πράγματα έχουν έτσι συμφωνούμε με τον εισηγητή ότι θα πρέπει να οικοδομήσουμε στο εφιστάμενο σύστημα που μας δίνει μια στέρεη βάση για τις μελλοντικέ εξελίξεις. Παρόλο αυτά υπάρχει ένα περιθώριο βελτίωσης. Η έκθεση παρουσιάζει ένα αριθμό προτάσεων ούτως ώστε να βελτιωθεί το σύστημα στα παρόντα όρια του. Η Επιτροπή χαιρετίζει την έφαση στη σημασία της αρχής εθνικής ανάθεσης. Ταυτόχρονα η έκθεση επισημαίνει μια αρνητική συνέπεια αυτής της αρχής. Τα υπάρχοντα ελλείμματα στη συμμετοχή των διαφόρων φορέων της κοινωνίας στον τομέα της υγείας και ασφάλειας, των ε, συμφερόντων των καταναλωτών, ε, ελλειπή συμμετοχή στη διαδικασία τυποποίησης. Η συμμετοχή αυτών των φορέων, των εκπροσώπων της κοινωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί προσδίδει στο σύστημα μια σημαντική πτυχή νομιμότητα και λογοδοσίας και βελτιώνει την ποιότητα, το επίπεδο της συνένεσης. Η Επιτροπή θα, θα εξερευνήσει συγκεκριμένου τρόπους ούτως ώστε να αυξήσει τη συμμετοχή των εκπροσώπων της ε, κοινωνίας ε, και ούτως ώστε να επιτευχθεί μια μεγαλύτερη ισορροπία στην διαδικασία αυτή εκπόνησης προτύπων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι σε σχέση με τον κεντρικό ρόλο των, της Αρχής της Εθνικής Ανάθεσης, ε, της ΕΝ και της ΕΝΕΛΕΚ, τα ευρωπαϊκά όργανα έχουν ένα ρόλο κλειδί στο ευρωπαϊκό μοντέλο τυποποίησης όλα τα εθνικά σώματα τυποποίηση θα πρέπει να παράσχουν μια στέρεη βάση για την δημιουργία μιας συνένεσης. Η έκθεση επισημαίνει κάποιες ε, διαφορές μεταξύ αυτών όσον αφορά τους σπόρους, την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και την δέσμευση των, των ενδιαφερόμενων στη διαδικασία τυποποίησης. Υπάρχει λοιπόν ένα περιθώριο βελτίωση στα επίπεδα των χωρών μελών. Παρόλο που το πρόβλημα της πρόσβασης στα πρότυπα δεν θα πρέπει να περιοριστεί ε, στο κόστος των προτύπων, η Επιτροπή χαιρετίζει την έκκληση των εθνικών φορέων να μειωθεί το κόστος ε, παρέχοντας κάποιες ε, δέσμες ε, τυποποίησης σε ένα χαμηλό κόστος και βελτιώνοντας την πρόσβαση ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η βεβαική τυποποίηση ε, έχει ένα σημαντικό δυναμικό για να υποστηρίξει τις δημόσιε πολιτικές. Εκτιμούμε ότι η έκθεση αναγνωρίζει αυτό το δυναμικό και τονίζει την ανάγκη να κινηθούμε προς νέες περιοχές ανάπτυξης προτύπων όπως είναι οι υπηρεσίες. Όπως επισημάθηκε από την έκθεση, το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο θα πρέπει να να συμβάλλει στην ευρωπαϊκή ε, καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την ιδιαίτερως ε, χρήσιμη και ε, έκθεση. Ευχαριστώ. Την πέμπτη στις 12 η ώρα. Η επόμενη συνεδρίαση θα διεξαχθεί αύριο 3η 19 Οκτωβρίου 2010 από τις 9 ως τις 30, από τις 15 ως τις 30, από τις 21 ως τις 24. Η μερίσια διάταξη έχει δημοσιευθεί και είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συνεδρίαση έριξε. Καλή νύχτα σε όλους. Thank you